αν κανείς δηλαδή μιλάει για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είτε στην Ευρώπη, είτε οπουδήποτε. Το Διεθνές Δίκαιο επιβεβαιώνει σαφώς ότι τα σύνορα δεν μπορεί να αλλάζουν με τη στρατιωτική δύναμη. Και αυτή είναι μια αρχή την οποία θα συνεχίσει να υποστηρίζει σταθερά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με ενωμένο τρόπο αυτή η ενότητα και η σαφήνεια μας έχουν καταστήσει Ε, τους στηρητές αρχής, μιας αρχής και μιας κατάστασης σε πολύ δύσκολες περιστάσεις. Η εικόνα που έχω στο μυαλό μου όταν σκέφτομαι τη Μέση Ανατολή είναι ότι δεν υπάρχει καμία διαδικασία. Δεν είναι ότι έχει σταματήσει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η ειρηνευτική διαδικασία. Η εικόνα που έχω στο μυαλό μου όταν ε, σκέφτομαι τη Μέση Ανατολή είναι, δεν ξέρω αν είναι αγγλική ή η έκφραση αυτή που χρησιμοποιώ, αλλά στα Ιταλικά αυτό λέμε, ότι κανείς ε, βάζει το πόδι του στην πόρτα ε, για να την εμποδίσει να κλείσει τελείω. Για να ξεκινήσει με όμως μια ερηνευτική διαδικασία που ε, θα βρει διεθνή συνένεση για τις παράμετρους, για την ανάγκη για την ύπαρξη μιας λύσης δύο κρατών. Θα χρειαστεί να υπάρξει πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές και από τη Washington. Από την ευρωπαϊκή πλευρά είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτό που όμως πρέπει να αποφύγουμε σήμερα μαζί με τους ε, συνεταίρους μας ε, στην περιοχή <clears throat> ιδιαίτερα με την Αίγυπτο, συνεργασία με την Αίγυπτο που έχει τόσο σημαντικό ρόλο για την αραβικό ε, ε, σύνδεσμο αλλά και για την Γάζα για να αποφύγουμε η τάση αυτή να συνεχιστεί να δεδρεωθεί και να καταστεί αναπότρεπτη σε βαθμό που όπως έλεγε η Έλενα η, η λύση των δύο κρατών να μην είναι πλέον δυνατή ώστε να αποφευχθεί η διάλυση αυτής της λύσης των δύο κρατών και να μην υπάρχει αδυναμία να επιτευχθεί όταν και εφόσον υπάρξει η πολιτική βούληση. Το ξέρω ότι είναι η προσέγγιση των ελαχίστων, αλλά πρέπει κανεί να είναι στην εξωτερική πολιτική. Ξημάμαι πάρα πολύ καλά την εντολή μου. Τη, τη θητεία μου την ξεκίνησα με την επίσκεψη στο Ισραήλ. Έλεγα τότε και μετά από 4,5 χρόνια λέω ότι αυτή η σύγκρουση μπορεί, μπορεί να λυθεί και, ξεκο... και είναι αλήθεια. Ακόμα το πιστεύω. Αλλά χωρίς την πολιτική βούληση των ενδιαφορεμένων μερών και χωρίς την διεθνή συνένεση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα όσον αφορά την λύση των δύο κρατών. Και εμεί οι Ευρωπαίοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν δεν είναι αυτή η λύση, δεν θα υπάρξει καμιά λύση. Και εντάξει, και το Ισραήλ δεν είναι και τόσο τέλειο. Ε, το ξέρει πάρα πολύ καλά και οι Παλαιστινοί το ξέρουν πάρα πολύ καλά σαν φίλοι της Παλαιστίνης, σαν φίλοι της περιοχής ολόκληρης. Ε, και να αναφερθώ και στην πρωτοβουλία του Αραβικού Συνδέσμου που εξακολουθώ να πιστεύω πως είναι καλή βάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπισμένη και θα συνεχίσει να είναι και σαφή σε αυτή την πεποίθηση πως είναι δηλαδή προς το συμφέρον των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων αλλά και ολόκληρη της περιοχής να συνεχιστεί η προσπάθεια για τον στόχο των δύο κρατών. Πρέπει αυτό να το πω ξεκάθαρα για όσους εδώ το ανέφεραν είναι πολύ ζωτικό και για την ασφάλεια των Ισραηλινών και του ίδιου του Ισραήλ. Αυτά είχα να πω νομίζω για αυτό το ζήτημα, κύριε Πρόεδρε. Και προσβλέπω στη συνέχιση της συζήτησής μας για το επόμενο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε. Είπατε εκπρόσωπε. Ολοκληρώνεται εδώ αυτή η συζήτηση και προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά την δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής ε, τη είπα τη προσώπου τη ε, Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, τη κυρία Φεντρίκα Μογκερίνη, για την κατάσταση στο Σουδάν. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο λαό του Σουδάν ζητεί αλλαγή. Τέσσερις μήνες τώρα είναι στους δρόμους, διαδηλώνουν. Μετά τις αυξήσεις ε, των τιμών στα βασικά αγαθά, αλλά ζητώντα πάνω απ' όλα ειρήνη και δικαιοσύνη. Η εικόνα μιας κοπέλας με λευκό φόρεμα που στεκόταν πάνω στην οροφή αμαξιού για να μιλήσει στον κόσμο έχει καταστεί συμβολική πλέον. Την κοπέλα αυτή την έχουν ήδη ονομάσει άγαλμα της ελευθερίας του Σουδάν. Και είναι προσδοκία του λαού η ελευθερία. Θέλει να επιτύχει ο λαός του Σουδάν. Θέλει αυτή η έκκληση για ελευθερία να εισακουστεί. Θέλει την αλλαγή ε, σε μια χώρα η οποία έχει υποφέρει τόσα. Την προηγούμενη εβδομάδα κατέλαβε την εξουσία ο στρατός, έθεσε τον Αλμπασίρ υπό κατοίκον περιορισμό. Ξέρετε ότι καταζητείται από διεθνή ε, δικαστήρια εγκλημάτων δικαίου και έχει στηθεί η έκδοσή του. Έχει ζητηθεί μια διετής μεταβατική περίοδος με στρατιωτικό συμβούλιο στην κυβέρνηση, αλλά που θα εκφράζει διαφορετικές τάσεις του στρατού, έτοιμα το οποίο και οι διαδηλωτέ, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμέσως απέρριψαν, ζητώντας εγγυήσεις για ταχύτερη μετάβαση σε πολιτική κυβέρνηση. Έτοιμα το οποίο και εμείς υποστηρίξαμε λέγοντας ότι ένα στρατιωτικό συμβούλιο δεν μπορεί να δώσει τις σωστές απαντήσεις στα αιτήματα των πολιτών και ζητώντας ταχεία και απρόσκοπτη μετάβαση σε πολιτική κυβέρνηση. Τις τελευταίες ημέρες ε, το στρατιωτικό καθεστώς προσπάθησε να καλύψει τις διαφορές επιδεικνύοντας ε, καλή βούληση άλλαξε η συνθέση Ιωτικού Συμβουλίου, επικεφαλής ε, της ε, υπηρεσίας πληροφοριών παρετήθηκε, κάποιοι από τους πολιτικούς κρατουμένους αποφυλακίστηκαν. Αυτό μπορεί να δείχνει ότι ίσως να υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις. Είναι σαφές πάντως ότι χωρίς γνήσια μετάβαση δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση στο Σουδάν έτσι. Πρέπει να αποτραπεί λοιπόν ένα σενάριο στρατιωτικής ε, διακυβέρνησης και να περάσουμε σε μια πολιτική διακυβέρνηση με γνήσια αποκάταση δημοκρατίας, με δημοκρατικές διαδικασίες, με ελευθερίες για να δώσουμε απαντήσεις στα αιτήματα των Σουδανών για πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι καταρχάς η αποτροπή της περαιτέρω βίας, η άρση της κατάπαυσης, ε, της απαγόρευσης κυκλοφορίας που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα του στρατιωτικού πραξικοπήματος και έκκληση να μην προβεί κανείς σε ε, προκλήσεις, καμία πλευρά. Επίσης ε, θα πρέπει οι μεταβατικές ε, αποφάσεις του Συμβουλίου, του πολιτικού Συμβουλίου, όπως αποφύλαξη των πολιτικών κρατουμένων και διαφύλαξη της ε, τάξης να υλοποιηθούν, πρέπει να καταδικαστεί κάθε εκτροπή που έχει εκδηλωθεί τους τελευταίους μήνες και έτσι να οικοδομηθεί ένα κλίμα κατάλληλο για πολιτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις έτσι ώστε όλες οι πλευρές και οι οργανώσεις των Σουδανών επαγγελματιών και οι πολιτικοί παράγοντες αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, του Συμβουλίου του Σουδάν να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Πράγμα κρίσιμο για την ε, συμφιλίωση και την ειρήνη σε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα προχωρώντας να επισημάνω ότι στην τελευταία μας διακήρυξη την προηγούμενη εβδομάδα για κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου της Επιτροπής Αφρικανικής Ένωσης, του κ. Μουσαφάκη, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω τα όσα είπε το Συμβούλιο Ασφαλείας και Ειρήνης Αφρικανικής Ένωσης ε, τις τελευταίες ημέρες, που ζητεί άμεση παράδοση της εξουσίας σε μια πολιτική αρχή μέσα στις επόμενες 15 μέρες, με μεταβατική περίοδο η οποία θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη μιας διαδικασίας διαβουλεύσεων βάσει της οποίας θα αναπτυχθούν οι όροι για τη μετάβαση σε ανώθευτες ε, και γνήσεις και ελεύθερες εκλογές. Όπως όλοι βεβαίως οι Σουδανοί θέλουμε αυτή η εκλογική αναμέτρηση να είναι στα χέρια των πολιτικών εκπροσώπων ε, και αυτό είναι το αίτημα στο οποίο και, το οποίο και εμείς προσυπογράφουμε όπως και πολλοί άλλοι. Όσο κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, όσο δεν έχει τη διαχείριση της μετάβασης η πολιτική εξουσία δεν μπορεί το η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει την νομιμότητα της μετάβασης του Στρατιωτικού Συμβουλίου. Μόλις όμως ε, παραδοθεί στα χέρια της πολιτικής εξουσίας η μετάβαση, τότε θα την παρακολουθήσουμε, θα τη συνοδεύσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους τόσο πολιτικούς όσο και οικονομικούς. Ευχαριστώ την υπατή εκπρόσωπο και τώρα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Τσέλερ έχει το λόγο. Στα πολωνικά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Για άλλη μια φορά λοιπόν η Αφρική, η Αλγερία τώρα και το Σουδάν έχουν ξεσπάσει σε συλλαλητήρια από πολίτες που ζητούν την, την από καθήλωση των δικτατόρων και το κατέφεραν, κατάφεραν. Ζητούν ε, ειρήνη, ζητούν ε, κοινωνίες στηριγμένες σε δημοκρατικές αρχές. Ξέρουμε όλοι βέβαια πόσο δύσκολο είναι ύστερα από τόσες δεκαετίες ε, βίαιης καταστολής και παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων στη χώρα και πάλι βλέπουμε ότι στο Σουδάν είναι πολύ ευάλωτη η κατάσταση. Κανείς δεν γνωρίζει αν είναι δυνατόν με βάση τις ερωτικές δομές που έχουν την εξουσία να γίνει η ομαλή μετάβαση προς, την πολιτική εξουσία. Πρέπει να αποκομίσουμε τα διδάγματα παρελθόντος και να ζητήσουμε με την Προεδρία της ΥΠΑ της εκπροσώπου και εκπροσώπευση όλων των κρατών σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση να πείσουμε τις ε, στρατιωτικές δυνάμεις του Σουδάν και να τις πείσουμε ε, για τη μετάβαση τους να μετατραπεί το Σουδάν σε μια νέα Λιβύη. Πρέπει οι πολιτικοί κρατούμενοι να αποφυλακιστούν. Οι μειονότητες που έχουν υποστεί καταστολή και καταπίεση πρέπει να αναγνωριστούν και να γνωστούν τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, τώρα ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Υπατεκπρόσωπε. Ελπίζουμε να υπάρξει αλλαγή που το απαιτεί ευρέως ο λαός του Σουδάν με επικεφαλής τις γυναίκες και ορισμένα τμήματα της κοινωνίας που είναι τα πιο προοδευτικά αυτής της χώρας. Αλλά το καθεστώς, το αυταρχικό καθεστώς υπάρχει εδώ και 30 χρόνια και σε αυτό προστίθεται και η ανθρωπιστική κρίση τεράστιων διαστάσεων. Γύρω στα 7 εκατομμύρια άτομα κινδυνεύουν από σοβαρό λοιμό στη χώρα αυτή. Ε, υπάρχουν γύρω στα 2 εκατομμύρια εσωτερικά μετατοπιστέντων και πάνω από 1 εκατομμύριο προσφύγων από γειτονικέ χώρες. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο όπου η Ερυθρέα, η Αιθιοπία, το Νότιο Σουδάν, η Σομαλία, το Τζιμπουτί. Επίσης, υφίστανται την πιο σημαντική ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο. Ένα σύνολο 20 εκατομμυρίων ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση άκρας ανάγκης. Και πρέπει να βοηθήσουμε αυτόν τον πληθυσμό μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά πάνω απ' όλα στηρίζοντας την ε, εγκαθίδρυση σταθερών καθεστώτων και της ειρήνης. Στηρίζω και στηρίζουμε ως ομάδα τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξέφρασε η πρόσωπος να στηρίξουμε μία μη στρατιωτική μετάβαση, να υπάρξει μία πολιτική κυβέρνηση και να προσπαθούμε να αποσταλεί ο Μπασίρ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να δοθεί πρόσβαση στους ε, γιατρούς και στους άλλους που χρειάζεται να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε από πλευρά τη Άλντε τώρα. Η κυρία Σχάκε, συνάδελφοι, η νεολαία του Σουδάν είναι ο λαός του Σουδάν. Η μέση ηλικία είναι 19 ετών και η νεολαία έκανε ακούστε τη φωνή της με την σαφή φωνή των ε, γυναικών ηγετών όπως η Άλλα Σάλα στην οποία αναφερθήκατε. Αυτοί είπαν αυτό και πέτυχαν μάλλον αυτό που δεν πέτυχε η διεθνή κοινότητα, την ανατροπή του Μπασίρ, ενό δικτάτορα, ο οποίο ε, είναι κατηγορούμενο ενώπιον του διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα, κατά του λαού του. Α θυμηθούμε πώ έχει κατάσταση. Η καταπίεση δεν μπορεί να καταπιέσει μέχρι τέλους τις εκκλήσεις για δημοκρατία και για αντιμετώπιση της διαφθοράς. Και οι σχέσεις με δικτάτορες για την βραχυπρόθεσμη μεταμετώπιση προβλημάτων όπως η μετανάστευση είναι κακή υπηρεσία προς τους νέους της Βόρειας Αφρικής και της Αφρικής γενικότερα. Και τρίτον, οι μεταβάσεις, οι μεταβατικές περίοδοι είναι πολύ ελπιδοφόρες αλλά και πολύ δυσχερείς διότι και οι θεσμοί και τα δημοκρατικά κινήματα και οι κοινωνίες των πολιτών προσπαθούν να βρουν τη σωστή λύση και οι πόροι του κράτους ε, απορροφώνται κυρίως από τις δυνάμεις καταστολής. Για να αποφύγουμε μια επανάληψη αυτών που συνέβησαν στην Λιβύη πρέπει να επενδύσουμε στη δημοκρατία και την ειρήνη ούτω ώστε ε, να μην καλύψουν το κενό οι διάφορες πολιτοφυλακέ που στρατολογούν απελπισμένους νέους. Κάποιοι είπαν από το Σουδάν ότι κόψαμε το κεφάλι αλλά το σώμα είναι ακόμη ζωντανό. Επειδή είναι η τελευταία συζήτηση που κάνουμε, κυρία εκπρόσωπε, σα ευχαριστώ Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη στον κόσμο, περισσότερο από ό,τι πριν από μια πενταετία. Σε εύχομαι κάθε περαιτέρω επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα για την κουα. η κυρία Βεζιά πολύ πριν να πω ότι μπορούσα και τι οφείλα να πω σε αυτή τη συζήτηση που η ε, ε, Ενωτική Ευρωπαϊκή Αριστερά ζήτησε για να στηρίξει τον λαό του Σουδάν, Κυρίω απέναντι σε αυτές τι χιλιάδε γυναίκες που διαδηλώνουν ειρηνικά ε, παρά την καταστολή, τις δεκάδε νεκρού και τι χιλιάδε συλλήψει. Συχνά είχα την ευκαιρία, ξέρετε κύριε Πατικπρόσωπε, να καταγγείλω εδώ τις σχέσει τη Ευρωπαϊκής Ένωσης με την δικτατορία του Ομάρα Αλμπασίρ. Αλλά δεν είναι πια και ε, τώρα η στιγμή. Είναι πολύ νωρί για να κρίνουμε το παρελθόν παρελθόν. Γι' αυτό θα πρέπει να περάσουμε πέρα από την ε, την απέτηση για πολιτική κυβέρνηση να βαρύνουμε ε, ώστε να πάμε προς μια μεταβατική κυβέρνηση. Η στρατηγική αυτή κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Ο αρχηγός ήταν ο υπεύθυνο του στρατού στην Ιεμένη και ο νούμερο 2 επίσης θα πρέπει και αυτοί να δικαστούν ε, μαζί με τον Ομάρ Αλμπασίρ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε αυτή τη χώρα. Μπορείτε να τους βοηθήσετε σε αυτό το αίτημα για αλλαγή καθεστώτος να μην μείνει μόνο μία επανάσταση χωρίς αποτελέσματα και από αυτό εξαρτάται η σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Νίνα Γκίλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε. Ακούσαμε ήδη ότι το Σουδάν έχει ε, αλλάξει πολύ. Ο, ο Μαρ ε, ε, ε, διώχθηκε μετά από 30 χρόνια δεν υπάρχουν ελεύθερα μέσα ε, και οι τιμές ε, των τροφίμων είναι ε, στα ύψη, όμως ο κόσμος και ιδιαίτερα οι γυναίκες του Σουδάν αντέχουν, είναι αθεκτικές και έχουν προσδοκίες και πραγματικά επιθυμούν αλλαγή. Σωστά υπάρχουν επιφυλάξεις για το στρατιωτικό καθεστώς. Πρέπει να υπάρξει μετάβραση προς μια πραγματική πολιτική κυβέρνηση μετά από ελεύθερες και διαφανείς εκλογές. Η Ένωση και εμείς θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη προς τους ειρηνικούς διαδηλωτές και θα πρέπει να μην επιτρέψουμε τη διετία ενός τέτοιου στρατιωτικού συμβουλίου να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είπατε εκπρόσωπε, εγώ καλωσορίζω τη δήλωσή σας ότι μόνο μια καθολική διαδικασία μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Σουδανών και να οδηγήσει σε πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα. Η ερώτησή μου όμως είναι ποιοι μηχανισμοί και συμμαχίες προτείνεται για να προχωρήσει η δημοκρατία βραχυπρόθεσμα και Επίση, η Υπηρεσία εξωτερική δράση εξετάσει στενά τι οικονομικέ ροές προ το Σουδάν, όπως έκαναν και οι ΙΠΑ όταν είδαν ότι ε, όταν μάλλον έβαλαν πρόστιμο στην BNP ε, Παρίμπας επειδή παραβίασε το ε, τις διατάξεις που ίσχυγαν για το Σουδάν. Ε, ε, θα εξασφαλίσετε ότι όλες αυτές οι διατάξεις το Διεθνέ Δίκαιο θα τηρηθούν πλήρως. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye με τον κύριο Μαριά πρώτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένα για το Σουδάν. Το τελευταίο διάστημα οι πάντες είχαν καταγγείλει την πολιτική του αλ μπασίρ και είχαν ζητήσει να πάρει μέτρα η ευρωπαϊκή ένωση προκειμένου να σταματήσει αυτή η κατάσταση να σταματήσει η καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να δοθεί ελευθερία στο σουδάν. τελικά όπως συμβαίνει πάντοτε ο ίδιος ο λαός δίνει τη λύση. γι' αυτό και με τις διαδηλώσεις κατάφερε καταρχάς να ανατρέψει τον αλ μπασίρ όμως οι δυνάμεις του καθεστώτος και κάποιοι άλλοι παραμένουν στην εξουσία μια και έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος. αυτή η στρατιωτική κυβέρνηση είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να περάσει στην δημοκρατική μετάβαση και είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να παραμείνει. γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη πίεση από πλευράς ευρωπαϊκής ένωσης ούτως ώστε να οργανωθούν δημοκρατικές εκλογές να μπορέσουν να λυθούν τα μεγάλα πολιτικά προβλήματα στο σουδάν και κατ' επέκταση τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα στη χώρα αλλά και τα ευρύτερα προβλήματα ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρόεδρε, ευχαριστώ. 30 χρόνια μετά είναι έτοιμο το Σουδάν, ετοιμάζεται μάλλον να γυρίσει σελίδα. Το αδύνατο γίνεται δυνατό. Ο Αλμπασίρ, δικτάτορας που καταστούνταν για χρόνια για τη γενοκτονία στον Ταρφούρ, ε, στις 11 Απριλίου, που, στις 11 Απριλίου καθερέθηκε. Ωστόσο, δεν σταμάτησαν οι κινητοποίησεις των πολιτών μετά την ανακατάληψη εξουσία από το στρατό. Εν της τη ε, διατύπωση διαμόρφωση στρατιωτική κυβέρνηση, έστω και προσωρινή, συνέχισαν οι πολίτε γιατί ανησυχούν ότι θα πέσουν και πάλι θύματα μια κατασταλτική κυβέρνηση όπω αυτή του Αλμπασίρ. Δεν θα σταματήσουν μέχρι ότου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσει του για την ελεύθερη μετάβαση και την ε, αποφυλάκηση των ε, αντιπολιτευμένων πολιτών, την αποκατάσταση τη ε, δημοκρατία και πάνω απ' όλα την εκαθάριση των μελών του προηγούμενου καθεστώτο του Αλμπασίρ. Έτσι λοιπόν μόνο μία διαδικασία αξιόπιστη με ανοιχτή προς όλους μπορεί να υποστηριχθεί από τον λαό του Σουδάν και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Χρειάζεται μια μετάβαση άμεση της εξουσίας σε μια πολιτική κυβέρνηση. Η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει πώς ε, ε, μπορεί να στηρίξει μια ειρηνική εξέλιξη και με οικονομικούς όρους. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αναγνωριστεί μια στρατιωτική κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χυθεί και άλλο αθώο αίμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παύλος Ρουμπίχη έχει τον λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πάνω απ' όλα για το Σουδάν, νομίζω είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και δεύτερον για μια ασφαλή το, ο δεύτερος στόχος είναι η ασφαλής και βιώσιμη ε, διατροφή. Στόχος 6, εκρίζωση των ασθενειών. Και σε αυτό θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να υλοποιήσουμε του στόχου. Ο έβδομο μεταξύ αυτών είναι οι ανανεώσιμε ε, πηγέ ενέργεια. Στην Ήπεθρο, λοιπόν, μαζί με τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, θα μπορούσαμε να καλύψουμε πάρα πολλέ από αυτέ τι ανάγκε για το μέλλον του Σουδάν, για τη σταθερότητα του Σουδάν, όπως άλλωστε και της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Dziękuję bardzo panu Rubikowi. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Και τώρα παρακαλώ την υπατή εκπρόσωπο να λάβει το λόγο. Thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τη σαφή στήριξη που έδωσαν στη θέση που υιοθετήσαμε, στη δουλειά που κάνουμε. Να απαντήσω μια ερώτηση, σε μια ερώτηση για τι στρατηγική και τι συμμαχίες θέλουμε να δημιουργήσουμε και ήδη δημιουργούμε για να πάει καλά αυτή η μετάβαση προς μια πολιτική, μη στρατιωτική κυβέρνηση και φυσικά ελεύθερες και έντιμες εκλογές. Όπως είπα και στην εισαγωγική μου παρουσίαση, παντού όταν συμφωνούμε, όπως συχνά συμφωνούμε, ο πρώτος συνομιλητής μας είναι η Αφρικανική Ένωση, που έλαβε σαφή θέση που νομίζω πως είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και το είπαν και ορισμένοι άλλοι συνάδελφοι. Αυτές οι αλλαγές στο Σουδάν είναι τμήμα μιας ε, βασικής, ε, μεγαλύτερης, ε, ριζικής αλλαγής της περιοχής γύρω από το κέρας της Αφρικής που είναι ελπιδοφόρα αλλά αντιμετωπίζει και προκλήσεις. Και σε άλλες χώρες της περιοχής Έχουμε νέε εξελίξει, για παράδειγμα, οι συνομιλίε μεταξύ Ερυθρέα και Αιθιοπία που ξεκίνησαν. Αλλά υπάρχουν σοβαρέ απειλέ ασφαλεία στην περιοχή. Με την πλήρη στήριξη και του δικού σα σώματο, και ξέρω ότι και το Συμβούλιο συμφωνεί θα προσπαθήσουμε να συνοδεύσουμε αυτή τη δημοκρατική μετάβαση ούτως ώστε να υπάρξει η δημιουργία μιας ε, πολιτικής κυβέρνησης και σε στενή συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και τις χώρες της ευρύτερη περιοχής να το επιτύχουμε αυτό, ιδιαίτερα οι γυναίκες και οι νέοι της Αφρικής ελπίζουμε να δουν τις προσδοκίες τους να υλοποιούνται. Αλλά όπως όλες οι μεταβάσεις η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Υπάρχουν ε, δυνατότητες αλλά και κίνδυνοι και προκλήσεις. Ευχαριστώ τους αδέλφους που ε, πήραν για τελευταία φορά το λόγο και με ευχαρίστησαν. Και θέλω και εγώ να τους ευχαριστήσω. Και για μένα ήταν ε, χαρά να συνεργάζομαι μαζί σας, ιδιαίτερα με τους αδέλφους που συμμετέχουν ε, περισσότερο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, αλλά θα είμαι εδώ μέχρι και την τελευταία συνεδρίαση, την πέμπτη για τις ψηφοφορίες, άρα θα έχουμε την ευκαιρία να ξανααποχαιρετήσουμε ένα τον άλλον και να ευχαριστήσουμε οι τους δε για την καλή συνεργασία τη τελευταία πενταετία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί εκπρόσωπε. Και εμείς είμαστε ευγνώμονες για τη δουλειά σας. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση και προχωρώ σε δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίω όσον αφορά τι διεθνεί απειλέ κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Καλωσορίζω με χαρά την ε, Υπουργό, κυρία Τσότ και τον ε, Επίτροπο κύριο Κίνγκ. Και Προεδρεύω πρέπει να σας πω με χαρά στο κομμάτι αυτό της συνεδρίασης, καθώς πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ιδιαίτερα με απασχολεί. Το έχω άλλωστε και στο χαρτοφυλάκι όμως μέλος του Προεδρείου, η εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ θα λάβουν χώρα τον επόμενο μήνα οι ευρωεκλογέ μέσα σε πολιτικά δεδομένα πολύ διαφορετικά από αυτά που είδαμε πριν από πέντε χρόνια. Είχαμε μαζικέ ε, ε, εκστρατείε παραπληροφόρηση και ε, παρισφρήσει στον κυβερνοχώρο με στόχο την απαξίωση και υπονόμευση των εκλογικών αναμετρήσεων στις χώρες μας αλλά και την πόλωση των κοινωνιών μας. Και ενώ εξελίσσονται εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε ένα τετραήμερο στα κράτη-μέλη, έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία και είναι αρκετά ευάλωτε σε επιθέσεις από τον κυβερνοχώρο. Κάποιες επιθέσεις που ενδεχομένως να αποδειχθούν επιτυχή σε ένα κράτος μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε εξελίξεις τύπου ντόμινο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν και ε, όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κινδυνεύουν να απαξιωθούν. Είναι απαραίτητο λοιπόν οι εθνικές αρχές, κρίσιμη περίοδος μάλιστα τώρα, αλλά όπως πάντα και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, προεδρική, εθνική, βουλευτική, τοπική, περιφερειακή που ε, θα αναπτυχθεί ε, στα κράτη-μέλη μέσα στην προσεχή περίοδο και μέχρι το 2020 να αντιμετωπίσει τις κυβερνοαπειλές. Εμείς έχουμε εντοπίσει την ανάγκη για μια συντονισμένη προσπάθεια προστασίας ελεύθερων γνήσεων και ανώθευτων δημοκρατικών ευρωπαϊκών εκλογών, ενίσχυση του δυναμικού μας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε απειλές και κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και την ενίσχυση της διαδικασίας της εκλογικής αναμέτρησης. Ένα θέμα το οποίο βλέπουμε να επανέρχεται τακτικά στο θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Συμβουλίου τους, επο... τους τελευταίους μήνες. Τα κράτη-μέλη αλλά και τα θεσμικά όργανα έχουν ρόλο σημαντικό και συμπληρωματικό στο πεδίο αρμοδιοτήτων του το καθένα να διαδραματίσουν προκειμένου να διαφυλάξουν τι δημοκρατικέ διαδικασίε. Χρειάζονται συντονισμένε προσπάθειε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κράτη-μέλη, αλλά και από την κοινωνία των πολιτών, αλλά και από τον κλάδο τη ηλεκτρονική επικοινωνία και τι διαγραμμικέ πλατφόρμε. Εστιάζουμε λοιπόν και πρέπει να εστιάσουμε τόσο στην εσωτερική όσο και στην εσωτερική, εξωτερική διάσταση τη απειλή αυτή στον κυβερνοχώρο. Στι 29 Μαρτίου θετήθηκαν συμπεράσματα από το Συμβούλιο για τη διεξαγωγή εγνήσεων ελεύθερων και δημοκρατικών ανώθευτων ε, ευρωεκλογών, μια νομοθετική πρόταση πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα που εντωμεταξύ είχε υιοθετηθεί από τους συνομοθέτες. Επίσης υπάρχει, είναι ευπρόσδεκτη ε, η πλατφόρμα για την κατάρριψη της παραπληροφόρησης και θα ήθελα κυρίες και κύριοι βουλευτές επί τη ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία η οποία επιτρέπει, επέτρεψε ταχύτατη υιοθέτηση των ε, κανόνων για την αποστολή ε, πολιτικών κομμάτων ή ιδρυμάτων και την ε, συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές. Μια συντονισμένη λοιπόν και ε, συμπεριληπτική προσέγγιση του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των επιθέσεων από τον κυβερνοχώρο και την παραπληροφόρηση αφορά τόσο το εσωτερικό στο και το εξωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απειλέ που να προερχόνται δηλαδή έξωθεν αλλά και από το εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να μην παραγνωρίσουμε κανένα κίνδυνο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε λύση, αλλά ταυτόχρονα να επιτρέψουμε τη συμμετοχή κάθε παράγοντα. Κάθε δράση λοιπόν που μπορεί να αναγνωρίζετε, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά. Ήδη κάποιε προτάσει ε, υιοθετήθηκαν τελευταίο μήνα. Η ε, Διεξαγωγή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ευρωεκλογών όπου μέλη της, ε, των εκλογικών επιτροπών των κρατών μελών εντοπίζουν απειλέ ε, και συντονίζουν τις προσπάθειές τους. Εθνικά σημεία επαφή για ταχύ ανταλλαγή πληροφοριών από εκστρατείε, παραπληροφόρηση επιδοκρατών μελών. Η ενίσχυση της στρατηγικής και τη επικοινωνίας, της επικοινωνιακής πολιτικής για τι αξίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα οικοσύστημα για τη διευκόλυνση των δικτύων ανεξάρτητων παραγόντων επαλήθευσης των ε, γεγονότων, ε, ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τον τρόπο χρήσης του διαδικτύου, βελτίωση των συνθήκων διεξαγωγής των εκλογών, συμμετοχή των διαφόρων παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών, η αξιολόγηση των κινδύνων και τα μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση τους μέσα από, ε, ώστε να προστατευτεί το εκλογικό σύστημα. Ένας κώδικας για την κυβερνοασφάλεια και την τεχνολογία των ψηφιακών εκλογικών αναμετρήσεων με την τάση με την προσπάθεια για την προστασία των ε, εκλογών του 2019 και μάλιστα έλαβε χώρα στους, ε, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από δύο εβδομάδες μόλις. Επίσης η ανάπτυξη της εκλογικής αναμέτρησης με βάση υπεύθυνη διαχείριση των διαγραμμικών δραστηριοτήτων, ένα, μια έκκληση για την πλήρη εφαρμογή ε, του κώδικα βέλτιστων πρακτικών και συνεργασία με τις αρμόδιες διεθνείς αρχές και υπηρεσίες. Όλα αυτά συμβάλλουν λοιπόν στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Η Προεδρία έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια χαρτογράφησης για τον εντοπισμό δράσεων και αντιμετώπιση του στο κατάλληλο επίπεδο και έτσι καταδεικνύει τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλουν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη για να καταπολεμήσουν τις προσπάθειες παραπληροφόρησης. Με τις αντιπροσωπείες μας ε, συνθέτουμε μια βάση για την αντιμετώπιση παραπληροφόρησης αλλά και την ανάπτυξη συζήτηση για περαιτέρω δράσεις και πέραν των εκλογών του 2019 που θα συζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε Επίτροπε Τζούλιαν Κίνγκ. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, όντως είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση και ευχαριστώ που την προγραμματίσατε γιατί ε, έρχονται γρήγορα, πλησιάζουν οι εκλογές και είμαστε σε τελευταίο στάδιο όσον αφορά τη λήψη μέτρων ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια αυτών των εκλογών. Τι έχουμε κάνει ε, κάποια πράγματα που κάνουμε τα έχετε ακούσει. Στους τελευταίους έξι μήνες περίπου έχουμε συγκεντρώσει τους επιτρόπους ε, εκλογών των κατορμελών, τους ειδικού για την ασφάλεια και για την προστασία των δεδομένων, ώστε να ε, ε, ενισχυθεί το δίκτυο για τη διοργάνωση των εκλογών, να μοιραστούμε τις καλύτερες πρακτικές, ώστε να ασφαλίσουμε με το δυνατό τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εκλογέ. Έχουμε καταστήσει ένα σύστημα γρήγορου συναγερμού ώστε να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε συντονισμένες πληροφορίες, εξατία συγγνώμη παραπληροφόρησης εδώ έχουμε έρθει σε επαφή με τις διάφορες ομάδες ώστε να ε, ενημερώσουμε για τη διαφάνεια των εκλογικών διαφημίσεων online. Έχουμε οργανώσει μάλιστα σεμινάριο μαζί σας, Πρόεδρε, στο Κοινοβούλιο για αυτό το σκοπό. Νωρίτερα αυτό το μήνα κάναμε συζητήσεις όσον αφορά την ασφάλεια μαζί με το Κοινοβούλιο, τα κράτη, ε, την, ε, τον Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ελέγξουμε πόσο ασφαλείς είμαστε ε, και αυτό ξεκίνησε με τον συνάδελφό σας, Αντιπρόεδρο Βίλαντ. Και είδαμε μεγάλες πλατφόρμες ε, του ίντερνετ που υπέγραψαν τις καλές πρακτικές για την παραπληροφόρηση πέρσι το ε, καλοκαίρι και ενισχύθηκε αυτό και με το πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης τον περασμένο Δεκέμβριο. Ε, οι πλατφόρμες αναφέρουν ε, κάθε μήνα το τι πρόοδο σημειώνουν για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, κυρίως της πολιτικής παραπληροφόρησης. Αναγνωρίζουμε ότι έχει υπάρξει όντως πρόοδος, αλλά οι εκθέσεις αυτές ή μάλλον οι αναφορές αυτές ήταν αποσπασματικές ε, και δείχνουν ότι σε κάποιου τομεί τουλάχιστον δεν γίνονται αρκετέ προσπάθειε. Κάποια αξιόπιστη πρόοδο έχει σημειωθεί στο τομέα των... της διαφάνειας των πολιτικών διαφημίσεων, ωστόσο οι πλατφόρμες πρέπει να βελτιώσουν την ανεξάρτητο έλεγχο για καλύτερη πρόσβαση για τους ελεγκτέ των στοιχείων, των... τους ειδικού και την κοινωνία των πολιτών. Δεν θέλουμε δηλαδή οι πλατφόρμες να αυτοβαθμολογούνται πρέπει να έχουμε πιο ταχεία και προφανή διόρθωση μέσω ας πούμε πιλωτικών προγραμμάτων για, όπως η πρωτοβουλία για τη διόρθωση των αρχείων όπως έχουν, έχει ξεκινήσει από την κοινωνία των πολιτών. Λάβαμε τις τελευταίες εκθέσεις των πλατφορμών για το τι κάνουν το Μάρτιο και θα δημοσιεύσουμε τη δική μας αξιολόγηση αυτών των αναφορών τις επόμενες μέρες. Κατά κάποιο τρόπο αυτό αντιπροσωπεύει μια τελευταία όφηση σε τομείς όπου μπορούμε ακόμα να επηρεάσουμε ρεαλιστικά στον καταπολέμηση της παραπληροφόρησης πριν από τις ευρωεκλογές. Εκ πρώτη όψεω, οι τελευταίε αναφορέ όντω ε, δείχνουν ότι έχει σημειωθεί και άλλη πρόοδο, για παράδειγμα όσον αφορά τη διαφάνεια για τι πολιτικέ διαφημίσει και τι διαφημίσει γενικότερα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια εκρεμή θέματα. Τέλος, να πω ότι τα κράτη-μέλη Έχουν ομάδες ε, ε, ανταπόκρισης για την ασφάλεια των υπολογιστών και θα συγκεντρωθούν για, σε ομάδα στα μέσα Μαΐου για την ασφάλεια των εκλογών και την ακαιρεότητα αυτών. Θα είναι τελευταία ευκαιρία για ένα έλεγχο για το πόσο ε, στεναρά είναι τα μέτρα ασφαλείας μας πριν τις ευρωεκλογές. Ένα ζήτημα που ήθελα να αναφέρω είναι ότι ένα από τα κρεμή ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τις πλατφόρμες και κυρίως με το Facebook πιο συγκεκριμένα είναι η απόφαση του Facebook να μην επιτρέψει διασυνοριακές πολιτικές διαφημίσεις. Ξέρω ότι αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες εδώ ε, στο Κοινοβούλιο. Όπως είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ανταλλαγή επιστολών με τον πρόεδρο Ταγιάννη, αυτή είναι μια απόφαση που έλαβε το Facebook. Δεν υπάρχει τίποτα στο κώδικα διοντολογία που περιορίζει τις πολιτικές διαφημίσεις μόνο στο χώρο, στο κράτος μέλος όπου ε, απευθύνεται η διαφήμιση. Ε, το θέμα είναι πώς θα γίνει η διαφήμιση και αλλού. Και έχει ληφθεί εξή απόφαση ε, και η ερμηνεία που δόθηκε στον σεβασμό των εθνικών εκλογικών νόμων έχει οδηγήσει σε ανησυχίες για το κατά πόσο οι θεσμοί ευρωπαϊκοί και τα ευρωπαϊκά κόμματα μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά πριν από τις ευρωεκλογές και το συζητήσαμε αυτό στη διάσκεψη των Προέδρων την περασμένη εβδομάδα και με χαρά μπορώ να σας πω τώρα ότι ο Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου και της Κομισιόν, οι γενικοί γραμματές δηλαδή, έχουν στείλει επιστολή στο Facebook όπου εκθέτουν πάλι τις ανησυχίες μας σαφέστατα και ζητούν από το Facebook να αναθεωρήσει τη θέση του σε αυτόν τον τομέα επιγόντως θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε αυτές τις προγραμματισμούς μας άμεσα με το Facebook σε μια επερχόμενη συνάντηση που έχουμε μαζί τους. Πρόεδρε, θέλω να πω ότι βέβαια το θέμα των ασφάλειας των εκλογών δεν πρόκειται να εξαφανιστεί μετά την 26η Μαΐου, γιατί όπως έχουμε ακούσει οι εκλογές συνεχίζονται, υπάρχουν εκλογές κάπου στην Ευρώπη κάθε εβδομάδα. Οπότε θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειές μας για να προστατεύουμε τις εκλογές και τις πολιτικές μας ζωές σε αυτήν την ψηφιακή εποχή. Θα γίνει σχετική συζήτηση τον Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια πρώτη αξιολόγηση για το πώς πήγαν οι ευρωεκλογέ και τι διδάγματα θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών επί τη βάση έκθεση ε, τη Προεδρία τη Επιτροπή και της του ΥΠΑ του εκπρόσωπου και θα μπορέσουμε έτσι να αποκομίσουμε διδάγματα και να θεσπίσουμε στρατηγικές για το μέλλον. Και ανάλογα με το τι θα συμβεί από σήμερα μέχρι τα τέλη Μαΐου, πιστεύω πως θα πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα αντιδράσουμε, πώς θα αποκομίσουμε όντως διδάγματα και πώς θα προβούμε στα απαραίτητα βήματα για το μέλλον. Επίσης θα αναθεωρήσουμε τον κώδικα διοντολογίας αργότερα ε, και θα ξανασκεφτούμε αν πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια γύρω από τις δραστηριότητες των online πλατφορμών στον πολιτικό ε, χώρο. Προσβλέπω λοιπόν στη σημερινή μας συζήτηση δεν είναι μια πρόκληση που θα μας απασχολήσει μόνο τις λίγες εβδομάδες που έρχονται, θα παραμείνει ως πρόκληση. Θα πρέπει να γίνουν ε, βέβαια δράσεις άμεσα τώρα εν ώψη των ευρωεκλογών, αλλά και στο μέλλον θα πρέπει να ε, ε, συνεχίσει να μας απασχολεί το θέμα, ώστε οι εκλογικές μας αναμετρήσεις να είναι όσο γίνεται πιο θωρακισμένες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επιτρόπε. Τώρα, ο πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Χιούμπνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, απτή δέσμευσή τους. Ε, για μας οι εκλογές είναι ένα κορυφαίο γεγονός της δημοκρατίας και αν ε, υπονομευθεί η κυβερνοασφάλεια των εκλογών μπορεί να χαθεί η εμπιστοσύνη στη δημοκρατική διαδικασία και στη δημοκρατική ηγεσία. Οι Ευρωπαίοι είναι όλο και πιο ευαισθητοποιημένοι και ανισχούν όλο και περισσότερο. Στα πρόσφατα, στα πρόσφατα ευρωβαρόμετρα λέγεται 61% ανησυχούν για την ενδεχόμενη προσπάθεια επηρεασμού των ευρωεκλογών μέσω του ίντερνετ για να μην αυτές οι απειλές και να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλέ το περιβάλλον διεξαγωγή των εκλογών, πρέπει να υπάρξει μια πλατιά προσέγγιση από όλη την κοινωνία και η διεθνή συνεργασία. Οπότε η τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για το καθεστώ και τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, ούτω ώστε να προστατευθεί η εκλογική διαδικασία από οποιαδήποτε επιγραμμική εκστρατεία παραλπροφόρηση που ε, βασίζεται σε κατάχρηση των προσωπικών του στοιχείων και εισαγωγή κυρώσεων για τους οργανισμούς που παραβιάζουν προστασία των δεδομένων ε, εσκεμένα για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρξει ένα ισχυρό πλαίσιο κυβερνοασφάλειας για να υπάρχει ευαισθητοποίηση σε επίπεδο κρατών μελών και στήριξη των κρατών μελών. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας να κάνουν τις πολιτικές τους επιλογές με δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από πλευράς των σοσιαλιστών, ο κύριος Κλοντ Μόρας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καλωσορίζω τα μέτρα που ανέλαβε ο Επίτροπος που εργάστηκε πολύ σκληρά για το θέμα αυτό. Αλλά είναι πολύ δυσχερές θέμα, συνάδελφοι. Η παρέμβαση στις εκλογές ε, συμβαίνει, έχει συμβεί και θα ξανασυμβεί. Και είναι επίγον το θέμα. Έκανε έκλειστο Κοινοβούλιο μέσω του κώδικα διοντολογία για να σταματήσει η διάδοση στο ίντερνετ των ψευδών ειδήσεων και θέλησε να υπάρξει αυτό ο κώδικας για την παραπληροφόρηση. Εξετάσαμε τι πρόοδος έχει σημειωθεί και είδαμε ότι το Facebook εξακολουθεί να έχει 160 εκατομμύρια από ψεύτικους χρήστες. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αν χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και δεν είναι μόνο το Facebook, είναι και το Google και το Twitter. Και ξέρουμε ότι και αυτοί έχουν υπογράψει λοιπόν αυτήν, ε, την, ε, αυτό τον κώδικα διοντολογίας. Πρέπει να αναλάβουμε δράσεις και στο ίντερνετ και εκτός. Στο ίντερνετ θέλουμε να υπάρχει πλήρης αλγοριθμική λογοδοσία και διαφάνεια. Είναι ουσιώδες, ούτω ώστε οι πολίτε να μπορούν να προστατεύονται από οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού του και να προστατευτούν οι εκλογέ από ξένε επεμβάσει και τα πολιτικά κόμματα και οι εκστρατείε θα πρέπει να δουν πώ χρησιμοποιούν τι κοινωνικέ πλατφόρμε για του εκλογικού σκοπού. Τώρα, στον πραγματικό κόσμο πρέπει να υπάρχουν εγγυήσει, κανόνε διαφάνεια για τη δαπάνη των πόρων, περίοδοι ε, ε, σκέψη χωρί εκλογική εκστρατεία και οι πλατφόρμε θα πρέπει να λένε ποιο περιεχόμενο ε, το προκαλείται από bots και να προσπαθούν να καταργήσουν τους ψεύτικους ε, χρήστες. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Αλλά επίση πρέπει να διασφαλίσουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι ο γενικό κανονισμό προστασία δεδομένων είναι ο μόνο τρόπο προστασία. Πρέπει να σταματήσει να είναι σε αδιέξοδο ο κανονισμό για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα, ιδιαίτερη προστασία των χρηστών κατά τη ε, στόχευση. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε για το Facebook και το σκάνδαλο τη εταιρεία Cambridge Analytica, αξιοποιώντα όλα τα μέσα που έχουμε στην Ένωση. Υπάρχουν τρει στον κόσμο που ρυθμίζουν την κατάσταση. Η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι εδώ, θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει στι ξένε δυνάμει που θέλουν να παρεμβαίνουν στι εκλογέ μα διαδικασίε. Δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα σημαντικότερο τώρα που επίκεινται ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Κλοντ, υπάρχει μπλε κάρτα από τον κύριο Έθεριτζ. Θέλετε να τη δεχτείτε. Το σκέφτομαι. Καλά, εντάξει. Παρακαλώ την ερώτησή σας. Ευχαριστώ, Κλόντ. Δεν θα είμαι επιθετικός. Σε ξέρω από τότε που είμαστε εδώ πέρα, είσαι λογικός άνθρωπος και δίκαιος. Δεν βλέπεις ότι παρά όλα αυτά τα οποία είπες στην ομιλία σου, πολλά τα κατανοώ και θα συμφωνούσα. Αλλά δεν κατανοείς και εσύ ότι υπάρχει κίνδυνος εάν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία από κρατικές αρχές ότι θα καταπνιγεί η ελεύθερη έκφραση. Ιδιαίτερα στο ίντερνετ. Διαφωνούμε σε πολλά, αλλά πάντα πιστεύω ότι έχεις κάθε δικαίωμα να πεις ό,τι πιστεύεις και αυτό πρέπει να ισχύει για όλους. Αυτό που είπα στην αρχή, ξέρω ότι θα συμφωνήσει και ο Επίτροπος όταν θα συνοψίσει τη συζήτηση. Δεν μιλάμε μόνο για την ελεύθερη έκφραση, που φυσικά είναι το πιο πολύτιμο δικαίωμα. Μιλάμε και για την παρέμβαση στις κυρίαρχες εκλογικές μας διαδικασίες από εξωτερικές ξένες δυνάμεις. Αυτό έχει αποδειχθεί στο 2016, στις προεδρικές εκλογές και στο δημοψήφισμα για τον Brexit. Δεν είναι ότι κάτι που πιστεύω. Έχει αποδειχθεί τεκμηριωμένα. Ελπίζω λοιπόν οι δημοκρατικές μας δομές να το αντιμετωπίσουν. Και τα θέματα όπως η ελευθερία έκφρασης και άλλα τόσο αγαπητά δικαιώματα υπονομεύονται από αυτές τις παρεμβάσεις. Ελπίζω και εγώ ότι καταλαβαίνεις ότι ε, εκτιμώ την ελευθερία έκφρασης όσο και εσύ, αλλά αν δεν υπάρχουν έλεγχοι στην παρέμβαση εναντίον αυτής, τότε ε, δεν επιτυχάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ για το ECR η κυρία Φωτίγα. Πρόεδρε, τεχνολογία της πληροφορίας και οι επιχειρήσεις επηρεασμού της κοινή γνώμης χρησιμοποιούνται εις βάρος της Δύσης από τη Ρωσία εδώ και καιρό και σε περιπτώσεις εκλογών. Γιατί, για να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη ε, την πίστη στη δημοκρατία για να οξύνουν οι φυστάμενους διχασμούς, ε, οι διαφωνίες, για να στρεβλώσουν την αλήθεια, για να ενισχύσουν ε, αφηγήματα φιλικά προς την Ρωσία. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε η τρίτη ανάγνωση στην Δούμα της ε, Ρωσίας ενός νομοθετήματος που απομονώνει το ρωσικό ίντερνετ από αυτό του υπόλοιπου κόσμου. Γιατί το ταχύτερο δυνατό πρέπει και για τη δική μας ασφάλεια αλλά και για την ασφάλεια των ε, ίδιων των Ρώσων πολιτών να μάθουμε το γιατί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα εκ μέρους της ομάδας ε, των φιλελευθέρων ο κύριος Τέλτσκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπατε και εσείς. Πολλά ήδη καλύφθηκαν, πολλά αληθινά πράγματα υπόθηκαν. Τα προσυπογράφω και πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε, έχουμε πραγματοποιήσει πρόοδο. Είπε όμως πολύ σωστά ο επίτροπο ότι ακόμα μένει να, πράξουν, να κάνουμε προόδου οπωσδήποτε. Αλλά α μην επαναλαμβάνω αυτά που υπόθηκαν και α θεωρήσω δεδομένα και σημαντικά τα όσα υπόθηκαν σε σχέση με τα όσα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Ας κοιτάξουμε και κάποιες άλλες πτυχές που πρέπει να γνωρίζουμε και ας ε, Κάνω και το παραλυσμό σε σχέση με τις πρόσφατες συνομιλίες και διαπραγματεύσεις για το νομοθέτημα για την κυβερνοασφάλεια που έχει μεγάλη σημασία για όλους μας ε, όσο έχει και η, υγεία και η ασφάλεια των πολιτών. Και αυτό που είπατε και εσείς ε, κύριε Υπουργέ, σημαντικό βεβαίω, αλλά δεν καταλαβαίνω, δεν βλέπω να το στηρίζουν ε, κάποια κράτη-μέλη με τις πράξεις τους. Δεν βλέπω να αναγνωρίζεται από μια ξηρά κρατών μελών πως όντως αντιμετωπίζουμε αυτή την απειλή στην οποία αναφέρθηκαν κάποιοι συνάδελφοι. Είτε πρόκειται για τις ευρωεκλογέ ή άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, τη ζωή, την ασφάλεια των πολιτών ή οτιδήποτε άλλο, ε, δεν βλέπουν ορισμένοι τους δουρίους ύπους που έχουν ε, παρισφρήσει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο δυστυχώ. Έτσι λοιπόν και παρά την πρόοδο σε επίπεδο νομοθετικό αλλά και σε όλα τα άλλα που αναφέρατε και εσείς σε σχέση με την ασφάλειά μας αλλά και σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Αυτό που χρειαζόμαστε και το γνωρίζει ο Επίτροπο ε, ω αυτό φρονώ, καθώ είχαμε τη συζήτηση πριν από μερικέ εβδομάδε, χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε να κάνουμε με έναν πόλεμο ο οποίος έχει εξαπολυθεί εναντίον μας όχι με όπλα πυροβόλα αλλά με άλλα όπλα διαφορετικού τύπου και πρέπει να τον αναγνωρίσουμε. Εάν δεν αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει αυτή η εμπόλεμη κατάσταση και αν δεν εστιάσουμε την προσοχή μας διαρκώς, όχι μόνο σε περίοδο ε, εκλογών, αλλά διαρκώς, τότε θα είμαστε πάντα ευάλωτοι και πάντα θα εφιστάμεθα επιθέσεις και ζημιά. Η κυρία Ματίας, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται όντως για ένα πρόβλημα πολύ περίπλοκο η παρέμβαση στις εκλογικές διαδικασίες και καταπολέμηση της, ε, τα καταπολεμά μάλλον κυβερνοασφάλεια, αλλά όχι μόνο αυτό, θα ήθελα να τονίσω κάποιες πτυχές που δεν αναφέρθηκαν. Εμείς υπερασπίζουμε το δικαίωμα στην ενημέρωση και υποστηρίζουμε τους δημοσιογράφους και τη δημοσιογραφία. Πρέπει να Ωστόσο, να αποφεύγουμε αυτούς τους χώρους όπου μπορεί ο καθένας να αναρτήσει οτιδήποτε θέλει, χωρίς καμία επαλήθευση ε, και αυτοί διαρκώς πολλαπλασιάζονται. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε τους εσωτερικούς ε, χειρισμούς και τη χειραγώγηση. Όμως άμα αν συνεχίζουμε να χειροκροτούμε τον κύριο Ζούκεμπεργκ για τους νέους κανόνες που ισχύουν στο Facebook, αλλά χωρίς ε, να κρίνουμε οτιδήποτε, τα πράγματα θα γίνουν πιο δύσκολα και χειρότερα για όσους ε, ασχολούνται με τις εκστρατείες. Χρειάζονται κατάλληλοι όροι αλλά και δράσεις που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση την ψηφιακή, με τη δημοσιογραφία και με τη μεγαλύτερη, περισσότερη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόχνερ. Ευχαριστώ πολύ. Εφόσον θέλουμε να προστατεύσουμε τις ελεύθερες ε, δίκες και μυστικές εκλογές στην ε, ψηφιακή μας εποχή, είμαστε ακόμη στα πρώτα βήματα. Καθυστερούμε και κάνουμε μόνο τα στοιχειώδη μέχρι τώρα. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αντιμετωπίζει επιτέλους αυτό το θέμα σοβαρά. Αλλά έχω ένα πρόβλημα για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις προσπάθειες επηρεασμού εκ των έξωθεν των εκλογών μας. Για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε τη συμφωνία για τη διτή χρήση. Ο κανονισμός για τη διτή χρήση μέχρι τώρα, εδώ και ένα χρόνο, εκρεμεί στο Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι οι εχθρικές προς την Ένωση δυνάμεις μπορούν πολύ εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στις τεχνολογίες μας, ούτως ε, ώστε, μεταξύ άλλων, να επηρεάσουν και τις εκλογικές μας διαδικασίες. Γι' αυτό κάνω επίγουσα παράκληση στο Συμβούλιο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Για το EFDD τώρα παρακαλώ, ο κύριος Έθεριτς. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να προστατευτούμε από αυτούς τους απέσιους Ρώσους που ελέγχουν το ίντερνετ, έτσι μας λέτε, ε? και στέλνουν παραπληροφόρηση, έτσι δεν είναι. Από μόνοι τους ε, κέρδισαν το δημοψήφισμα για τον Brexit, ε, γιατί έχουν πολλά bot. Αλλά δεν ανησυχούμε καθόλου για το γεγονός ότι αυτό που θα μπορούσε να οδηγήσει στη λογοκρισία και στον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης. Είναι θέμα εξουσίας. Η εξουσία των καταστημένων δυνάμεων μέσω των ε, κύριων μέσων ενημέρωσης είναι πρωτόγνωρη. Κοιτάξτε το BBC που είναι ο μεγαλύτερος ε, πάροχος περιεχομένου στο ίντερνετ. Είναι κυρίως ε, υπέρ του κράτους. Αυτό δεν σας πειράζει γιατί δεν είναι το κράτος κατά της Ένωσης. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Φυσικά το Facebook και άλλες πλατφόρμες πρέπει να βρίσκουν τα bot και να τα διαγράφουν. Αλλά αν δώσετε τόση εξουσία στο κράτος για να κλείσει ό,τι γουστάρει, ποιος θα το κάνει. Για φανταστείτε. Φανταστείτε. Εάν ένας ε, κεντροδεξιός ε, που είναι υπέρ του καπιταλισμού και κατά των πρασίνων είχε την εξουσία στην Ένωση, θα ήταν τρομερό αυτό, ε και ξαφνικά παρεμποδίσουν την ελεύθερη έκφραση στο ίντερνετ όσων διαμαρτύρονται κάτω των ιδεών του. Πώ θα το βλέπατε αυτό, Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Α αφήσουμε στου ανθρώπου το δικαίωμα να εκφράζονται. Μα λέτε για ελευθερίε εδώ μέσα. Ποια ελευθερία είναι πιο σημαντική από την ελευθερία τη έκφραση, την ελευθερία λόγου. Κατά τη γνώμη μου. Το πιο σημαντικό είναι αυτή η ελευθερία. Η περισσότεροι εδώ μέσα είναι άνθρωποι με τους οποίους διαφωνώ, αλλά θα ήμουν πρώτο στα οδοφράγματα για να περασπιστώ το δικαίωμά σας να εκφράσετε τις απόψεις σας όπως και αν θέλετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Έθεριτς. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον Πάβελ Τελίτσκα. Ναι, παρακαλώ, Πάβελ. Ευχαριστώ πολύ που δέχεστε την ερώτησή μου. Συμφωνώ για την ελευθερία έκφρασης αλλά στις παρατηρήσεις σας δεν άκουσα καμία ανησυχία για τις ενδεχόμενες επιθέσεις από την Ανατολή ή από αλλού και παρέμβαση στις ευρωεκλογέ. Οπότε ερώτηση. Συμμερίζεστε αυτή την ανησυχία. Και αν ναι, πώς θα την αντιμετωπίσετε αυτή την απειλή. Πώς θα ε, προσπαθήσετε να μειώσετε τον κίνδυνο. Ο κύριος Έθεριτς. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, πολύ σκόπιμη. Βεβαίω, συμμερίζουμε αυτή την ανησυχία. Δεν θέλω κανεί να παρεμβαίνει στι ελεύθερε εκλογέ μα. Αλλά, αν έχω να επιλέξω. Γιατί κοιτάξτε, η ζωή είναι όλα αποφάσει. Εάν η επιλογή είναι από τη μία να απαγορεύσω να εκφράζονται ελεύθεροι άνθρωποι και τον κίνδυνο το κράτος να κυλήσει προς τον ολοκληρωτισμό, προτιμώ τους κινδύνους από την ελεύθερη έκφραση αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε την παρέμβαση ξένων υπηρεσιών στις εκλογές μας. Σας ευχαριστώ. Ένφ, κύριος Μπάτν είναι εδώ. Όχι από ό,τι βλέπω. Επομένως θα παρακαλέσω τον κύριο Λεπέν να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν από 25 χρόνια από αυτό το βήμα ο Φρανσουά Μιτερό είπε μία φράση λακωνική αλλά ανακριβή εθνικισμός ίσον πόλεμος έντονη εικόνα, ισχυρή εικόνα αλλά λάθος μήνυμα ο εθνικισμός τότε μπορεί να ήταν εθνικές ε, Εθνική στρατή. Τώρα δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι τα στρατεύματα του πολικού Βλαδιβοστόκ είναι ένας, ε, μια απειλή ε, τεκτονικού χαρακτήρα για την Ευρώπη. Εδώ έχουμε ακόμα περισσότερα μια μεγάλη απειλή για την ανεξαρτησία τις ελευθερίες, την επιβίωσή μας. Έχουμε καθήκον υποχρέωση να τις αντιμετωπίσουμε για να καταστήλουμε την απειλή αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, σήμερα δεν είναι παρακέλυφος και είναι μια, ε, ένας ε, μία μέγενη η οποία εμποδίζει την ε, δράση των πολιτών και των εθνών δεν τους επιτρέπει κανένα περιθώριο. Ό,τι και να λένε φεντεραλιστές ε, δεν υπάρχουν ούτε ευρωπαϊκά έθνη ούτε λαοί ευρωπαϊκοί. Το ίδιο αυτό το σώμα στο οποίο συμμετέχετε εσείς εκλέγεται από τα έθνη που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έθνος είναι το πολιτικό, ηθικό ε, στοιχείο, η ραχοκοκαλιά του κάθε κράτους και όλων των διεθνών οργανισμών όπως των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι λοιπόν είναι το πλαίσιο το πιο φυσιολογικό και αποτελεσματικό το έθνος για να επιτρέπει να ζουν και να ευημερούν οι λαοί ε, που συμμετέχουν σε αυτό με την αγάπη στην πατρίδα, στο έδαφος, στην ιστορία. Η ε, πατρίδα είναι αυτή που ξεπερνά και παρατείνει το πεπρωμένο του καθενός. Είναι αυτή η οποία εγγυάται το μέλλον της κάθε γενεάς. Υπάρχει βεβαίως ένας ευρωπαϊκός πολιτισμός, ένας απαυγάζων ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο οποίος απαιτεί την στενή συνεργασία των εθνικών κρατών, των εθνών, των κρατών όλης της Ευρωπαϊκής Υπήρου και όχι μόνο της Δυτικής Ευρώπης. Έτσι λοιπόν από τα 3 στα 8 δισεκατομμύρια πολίτες στην οικουμένη με την γεωμετρική πρόοδο της αύξησης της δημογραφικής και το μεγάλο κίνδυνο της μεταναστευτικής απειλής της οποίας μόνο την ε, σκιά μπορούμε να δούμε ακόμα Απειλεί λοιπόν την Ευρώπη αυτή, την ε, υπηρετική αυτή Ευρώπη που έχει δημογραφικό έλλειμμα και είναι υποχρεωμένη να βρει μια ισορροπία μεταξύ των αναγκών και της παραγωγής του κόσμου, μεταξύ της εξαθλίωσης στον κόσμο, της φτώχειας ε, που καθιστά την Ευρώπη ένα Ελντοράντο, μια γη της επαγγελίας, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πρόσωπο της μέδουσας που θα μας κάνει παρά το πρόσωπο της ε, ε, σχεδίας μέδουσα που θα μας κάνει να βυθιστούμε όλοι να βαγεί στον ωκεανό. Και πρέπει πάνω απ' όλα να γνωρίσουμε τους λαούς που απαρτίζουν την Ευρώπη. Εσείς βουλευτές που μείνατε τυφλοί, τα τότα των τενούν, τα τόματα θα είσαστε μπροστά στο μέλλον σας υπόλογοι.